Καλημέρα και ειδικά στον αγαπητό συνάδελφο Όγγεν Φρόιντ. Καλημέρα και σε όλους. Θα συνεχίσω βέβαια στα αγγλικά διότι τα χαρτιά και σημειώσεις μου είναι στη γλώσσα αυτή. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα, αγαπητοί συνάδελφοι, συνεχίζουμε με το σημείο 12 της ημερήσιας διάταξης με ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τους κινδύνους ασφαλείας από τα καταβυθισμένα πολεμοφόδια. Μας υπενθυμίζουν οι κατά καιρούς ότι υπάρχουν όντως καταβυθισμένα πολεμοφόδια στον βυθό της θάλασσας, ε, θαμένα όταν εκρήγνεται σε, πολεμικές, σε πρώην εμπόλεμες ζώνες. Ε, πολλές φορές ε, ψαράδες δηλητηριάζονται από διάφορα αέρια που εκλείονται από πολεμοφόδια θαμμένα από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Εκατό χρόνια αργότερα. Σήμερα λοιπόν θα συζητήσουμε για αυτά τα χημικά όπλα και τα κατάλοιπά τους, τα οποία αποτελούν απειλή για την θαλάσσια ζωή, για τους παράκτιους ε, πληθυσμούς και για τον βυθό της θάλασσας. Θα γίνει ανταλλαγή απόψεων με προσκεκλημένου στην Εντόρα Μπαρέιρα Ράμπο, αρμόδια πολιτική τη μονάδα Α3, στρατηγικέ για τι θαλάσσιε λεκάνε, θαλάσσια περιφερειακή συνεργασία και ασφάλεια στην θάλασσα από την Γαμαδέλτα Μάρε. Καλώ ήρθατε. Και από τον Πιέρ Φραντσέσκο Μωρέτη επιστημονικό σύμβουλο από την Πρωτοβουλία Κοινού Προγραμματισμού Οκεανή του Εθνικού Συμβουλίου Ερευνών της Ιταλίας. Θα δώσω πρώτα το λόγο στην κυρία Μπαρέιρα Ράμος και έπειτα στον κύριο Μωράτη. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σε όλους. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω φυσικά για την σημερινή πρόσκληση. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι σήμερα εδώ για να σας παρουσιάσω αυτό το τόσο σημαντικό θέμα των βυθισμένων, καταβυθισμένων πολεμοφοδίων. Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στο θέμα αυτό, στα καταβυθισμένα πολεμοφόδια και άλλο πολεμικό υλικό που απορρίπτεται στην θάλασσα. Είναι σημαντικό πρόβλημα σε όλο τον κόσμο και στην Ευρώπη. Το θέμα αυτό είναι ιδιαίτερα ορατό στην Αδριατική, τη Βαλτική και περίπου 4.000 τόνοι χημικών πολεμοφοδίων βυθίστηκαν στη Βαλτική μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι αριθμοί λοιπόν είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακοί. Όμως πρέπει να δώσουμε σημασία σε όλες τις ε, διαφορετικές διαστάσεις του προβλήματος. Τα πολεμοφόδια στη θάλασσα καταρχάς αποτελούν κίνδυνο για την ασφάλεια και το περιβάλλον. Οι κίνδυνοι αυτοί γιγαντώνονται από το γεγονός ότι τα πολεμοφόδια αυτά περιέχουν χημικά, ε, θείο, αέριο μουστάρδας και άλλα επικίνδυνα χημικά και αποτελούν ενδεχόμενες απειλές για τα θαλάσσια οικοσυστήματα αλλά και για την ανθρώπινη υγεία. Κατόπιν τούτου θα ήθελα να, επι... να τονίσω επίσης ότι τα πολεμοφόδια εφόσον εκραγούν και αν εκραγούν αποτελούν εμπόδιο στην οικονομική ανάπτυξη. Η αυξανόμενη χρήση του βυθού της θάλασσας, για παράδειγμα, για την ε, διέλευση υπόγειων αγωγών ή ε, άλλων ε, σταθμών ε, παραγωγής ενέργειας είναι κάτι που επηρεάζεται πάρα πολύ από αυτά τα πολεμοφόδια. Πολλές φορές ολόκληρες ε, περιοχές επίσης είναι απαγορευμένες για τους ψαράδες ακριβώς επειδή η αλίευση είναι πάρα πολύ επικίνδυνη λόγω των καταβυθισμένων πολεμοφοδίων. Χρειάζεται λοιπόν ειδικό σχεδιασμός για την θάλασσα έτσι ώστε να αποτραπεί ο κίνδυνος ε, από τα πολεμοφόδια αυτά. Χρειάζεται λοιπόν να χαραχθεί στρατηγική ανταπόκριση στο πρόβλημα αυτό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε δώσει έμφαση στο εθνικό και περιφερειακό επίπεδο για τον έλεγχο και τον καθαρισμό των ε, τοποθεσιών αυτών από τα καταβυθισμένα πολεμοφόδια. Επίσης όμως πρέπει να συνεισφέρουμε και με την έβρεση λύσεων για την ε, πρόκληση αυτή. Κατανοούμε λοιπόν ότι η χαρτογράφηση και ο έλεγχος των περιοχών όπου βρίσκονται τα πολυμοφόδια είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο. Υπάρχει ένα δίκτυο AMONET το οποίο παρατη... κάνει έλεγχο και λειτουργεί ως παρατηρητήριο και καταγράφει τις ε, τοποθεσίες και διάφορα στοιχεία για τα πολεμοφόδια για τον ε, βορειοανατολικό Ατλαντικό καθώς ε, επίσης υπάρχει συνεργασία με εθνικά υπουργεία αλλά και με τα Ηνωμένα Έθνη. Χρειάζεται να ληφθούν σοβαρά οι κίνδυνοι για την ασφάλεια και γι' αυτό χρειάζεται μια συντονισμένη απάντηση αυτό αναφέρεται στο σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το οποίο εγκρίθηκε το 2014 από το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων και αναθεωρήθηκε το 2018. Το σχέδιο δράση λοιπόν για την ασφάλεια στη θάλασσα αναφέρει τις προθέσεις μας για την ε, περισυλλογή και εξουδετέρωση των καταβυθισμένων πολεμοφοδίων μέσω μίας ενιαίας συντονισμένης απάντησης. Επίσης, Αξίζει να σημειωθεί ότι το σχέδιο δράσης Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενίσχυση της ασφάλειας αναφέρει επίσης τον κίνδυνο από ενδεχόμενες εκρήξεις πολεμοφοδίων. Τον Ιούνιο του 2007 ε, η έκθεση για την ασφάλεια τόνισε την ε, σημασία της συνεργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισμών όπως τα Ηνωμένα Έθνη και όχι μόνο, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον ε, τομέα αυτών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεισέφερε στο ψήφισμα Α71 των Ηνωμένων Εθνών για το ίδιο θέμα. Οι συμβάσεις, οι περιφερειακές συμβάσεις για θαλάσσια ζητήματα επίσης είναι πολύ σημαντικές διότι θα αυξήσουν τις συνέργειες μεταξύ κρατών και επίσης θα οδηγήσουν στην ε, ανάπτυξη διάφορων έργων διακρατικών ακριβώς για τον ε, σκοπό αυτό. Ιδιαίτερα στην ε, περιοχή της Βαλτικής υπάρχει και η αντίστοιχη στρατηγική που περιέχει τέτοιες ε, διατάξεις. Επίσης, έχουν γίνει προτάσεις για διάφορα έργα υπό το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, τα οποία θα προωθήσουν την ε, γαλάζια οικονομία. στο πρόγραμμα αυτό θα στηριχθούν καινοτόμε λύσεις οι οποίες θα εντοπίσουν τα καταβυθισμένα πολυμοφόδια και θα ε, οδηγήσουν στην περισυλλογή τους. Χρειάζεται λοιπόν επίσης να προσθεθεί το θέμα αυτό και στην ε, ατζέντα για την θάλασσα, το, η οποία θα η οποία παρουσιάστηκε μάλλον σε συνδυασμό ε, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ε, τους ε, εθνικούς φορείς. Έτσι θα αυξηθούν οι συνέργειες και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βρίσκεται σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. μια, θα διοργανώσει μάλλον μια εκδήλωση για το θέμα αυτό στις 20 Φεβρουαρίου στις Βρυξέλλες. Και φυσικά θα είμαστε σε επαφή με τη γραμματεία της ε, Επιτροπής σας ε, και θα παρέχουμε όλες τις ε, λεπτομέρειες σχετικά. Έχουμε επίσης στείλει πρόσκληση στην κυρία Φωτίγκα, πρόεδρο της Επιτροπής ΣΕΝΤΕ, η οποία θα μιλήσει στην εκδήλωση αυτή, ελπίζουμε, αλλά και τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής είναι φυσικά ευπρόσδεκτα στην εκδήλωση αυτή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν για να δούμε τις προκλήσεις που υπάρχουν για το θέμα αυτό. Θα, η εκδήλωση θα έχει ομιλίε από ε, εμπειρογνώμονε και θα συζητηθούν οι πιθανές λύσεις σε αυτό το πολύ σημαντικό πρόβλημα, αυτή τη σημαντική απειλή για την ασφάλεια και την υγεία. Σας ευχαριστώ. Thank you very much for... Ευχαριστώ Και τώρα ο κύριος Μωρέτη έχει το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ το Κοινοβούλιο που κάλεσε το Εθνικό Συμβούλιο Ερευνών της Ιταλίας ε, που ασχολείται με τους ωκεανούς. Ε, θα ήθελα να μιλήσω Ιταλικά, ε, συγγνώμη, ε, Αγγλικά, παρότι είμαι Ιταλός γιατί εκπροσωπώ 28 κράτη-μέλη. Θα ήθελα να σας δώσω κάποιες εξηγήσεις για αυτή την πλατφόρμα, η οποία ξεκίνησε να λειτουργεί το 2011 από το Συμβούλιο ε, για να αντιμετωπίσουμε τις παγκόσμιες προκλήσεις γιατί δεν μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε μεμονωμένα κάθε κάθε μελος ε, Κανένα Κάνα κράτος-μέλος δεν μπορεί από μόνο του να βρει λύσεις στι παγκόσμιες αυτέ προκλήσεις οι συμμετέχουσες χώρες και το Συμβούλιο ε, συνένωσαν τις προσπάθειές τους για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις. Και αυτό το θέμα ε, στους ωκεανούς ε, είναι μεγάλο πρόβλημα. Έχουμε 21 χώρες που συμμετέχουν, συν την Κομισιόν που είναι παρατηρητής και θα... Θέλαμε να πούμε ότι δεν κάνουμε μόνο συνεργασία με τα Υπουργεία Έρευνας και Καινοτομίας, αλλά το Αλίας, ε, των Μεταφορών, το Υπουργείο Ανάπτυξης, ε, τα Υπουργεία μάλλον Ανάπτυξης διαφορών χωρών. Ε, και χάρη σε αυτές τις πρωτοβουλίες βλέπουμε πώς η έρευνα και η καινοτομία μπορεί να συνεισφέρει για να επιληθούν οι προκλήσεις. Άλλες πρωτοβουλίες που προωθούμε είναι μια μακροπρόθεσμη θεώρηση με τα Υπουργεία, δέσμευση δηλαδή υπάρχει σε υψηλό επίπεδο και χρησιμοποιούμε τη λεγόμενη μεταβλητή γεωμετρία. Ε, δεν είναι ότι συμφωνούμε όλοι στις ίδιες δράσεις. Υπάρχει πρόκληση μπροστά μας και ο στόχος είναι να πετύχουμε την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Όταν εσύ όμως θες να εφαρμόσεις μια δράση, κάνεις αυτό που νομίζω ότι είναι σημαντικό στο δικό σου επίπεδο. Και αυτή είναι η καινοτομία στο τρόπο συνεργασίας δηλαδή των κρατών μελών. Έπειτα, ως συνήθως, στην Ευρώπη έχουμε ε, την, ε, το θεματολόγιο για τη στρατηγική έρευνα και καινοτομία. Είναι ένα πλαίσιο, φανταστείτε. Είναι αδύνατον ουσιαστικά να αντιμετωπίσουμε όλες ε, τις πτυχές μαζί. Είναι ένα μενού, έτσι. Αλλά έχουμε μέσα σε αυτό το μενού δέκα δραστηριότητες ή ε, προτεραιότητες αλλά όπως είπα και πριν εστιαζόμαστε σε κάτι που είναι σημαντικό για μας, που βοηθάει στην αντιμετώπιση του προβλήματος, που είναι οριζόντιου χαρακτήρα. Προσπαθούμε δηλαδή να έχουμε διαφορετικές δράσεις στην Ευρώπη και καινοτόμε. Δεν θέλουμε να εστιάσουμε σε ένα μόνο πρόβλημα, αλλά σε δράσεις που πραγματικά μετασχηματίζουν τον τρόπο που η έρευνα βρίσκει λύσεις. Ε, ένα από τα θέματα είναι τα πολυμοφόδια στη θάλασσα που μας απασχολούν δηλαδή. Ε, όπως είπε και τώρα, έχουμε αυτά τα πολεμοφόδια στη θάλασσα, ε, δεν τα ξέρουν όλοι ίσως, αλλά η ιδέα ποια είναι. Ε, ε, θεωρείται χαμηλού κινδύνου αυτό το πρόβλημα. Δεν θεωρούμε ότι θα εκραγούν κατά ανάγκη όλα αυτά τα πολεμοφόδια, ας το πω έτσι. Έχουμε την εξή ιδέα έχουμε πολεμοφόδια τα οποία δεν αντιμετωπίζουν, δεν μας ε, ε, δημιουργούν μεγάλους κινδύνους ε, σε ό,τι αφορά την πιθανότητα έκρηξης, αλλά έχουμε και την, το πρόβλημα της διαρροής στη θάλασσα. Λοιπόν, εμείς ως ερευνητές δεν θέλουμε με τις πρωτοβουλίες αυτές, τις ερευνητικές, να αφήσουμε αυτά τα πολεμοφόδια να εκραγούν. Το θέμα αυτό δεν είναι μόνο θέμα κατεπήγοντος, ας γιατί μπορεί να κρακούν αυτά τα πολεμοφόδια. Το θέμα είναι και θέμα χώρου που καταλαμβάνουν στους ωκεανούς. Ε, όλο και περισσότερο καταλαμβάνουν χώρο, ε, όγκο στο, στον ωκεανό και δεν το θέλουμε αυτό. Τι κάνουμε λοιπόν. Στην αρχή είπαμε ότι αυτό το πρόβλημα θέλουμε να το αντιμετωπίσουμε. Ε, δεν μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε όλα τα προβλήματα, αλλά αυτό μπορούμε. Ε, όμω ότι τελικά ε, σε κάποια Υπουργεία, όχι στο Υπουργείο Άμυνα, ε, λέγανε ότι κοιτάξτε, αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να το σκεφτούμε. Ξοδέψαμε ένα χρόνο λοιπόν για να καταλάβουμε αν υπήρχε πραγματικά ε, δυνατότητα να συνεισφέρει η ερευνητική κοινότητα στο πρόβλημα και στην αντιμετώπιση του. Προσπαθήσαμε λοιπόν να στείλουμε τελείως ε, διαφορετικό μήνυμα. Είπαμε, εντάξει θέλουμε να προλάβουμε τα κατεπήγοντα, δεν θέλουμε να συμβούν και να δημιουργηθούν κατεπήγουσες καταστάσεις, θέλουμε να τις αντιμετωπίσουμε και να τις προλάβουμε. Ε, υπάρχει το θέμα της ασφάλειας, safety. Αυτό μπορούμε να το πουλήσουμε εύκολα. Θέλουμε να υποστηρίξουμε την, τους νομοθέτες ε, για να, και να πλαισιώσουμε τον τρόπο που παρεμβαίνουν και νομοθετούν. Ε, θα πρέπει όμως να βρούμε και νέες λύσεις ε, ε σε ερευνητικό επίπεδο. Συχνά ο στρατός ή το στρατιωτικό επίπεδο αντιμετωπίζει αυτό το θέμα και το ΝΑΤΟ βέβαια. Ε, χρειαζόμαστε χρόνο για να εισαγάγουμε διαδικασίες. Γι' αυτό λοιπόν θέλουμε να ψάξουμε να βρούμε ε, το πώς σκέφτονται, τι, τι λύσεις έχουν να προτείνουν διάφοροι τομείς, ε, τα διάφορα επίπεδα. Ε, η ερευνητική κοινότητα αλλά και άλλες κοινότητες. Ε, στις αρχές θεωρούσαμε ότι βλέπαμε μάλλον την, ε, πολλοί βλέπουν την ερευνητική κοινότητα σαν εντελώ ανεξάρτητη. Δεν είναι σωστό αυτό. Ε, Εμεί τι κάναμε, θέλαμε μια συνολική σφαιρική προσέγγιση. Αμέσω λοιπόν ενημερώσαμε το ΝΑΤΟ. Ε, είμαστε στην Ευρώπη και όλες ε, και οι περισσότερες τεχνολογίες που χρησιμοποιούμε ε, είναι τεχνολογίες που χρησιμοποιεί και, ο ΝΑΤΟ, και το ΝΑΤΟ. Ε, υπήρχαν ομάδες μέσα στο ΝΑΤΟ που απασχολούνταν ήδη με αυτό το θέμα. Αρχίσαμε λοιπόν να ανταλλάσσουμε πληροφορίε. Ε, τους καλέσαμε και σε κάποιες ε, έτσι, προσπάθειες που κάναμε στην αρχή στην Πορτογαλία. Ε, προσπαθήσαμε να γεφυρώσουμε τις διάφορες κοινότητες. και τους κοιτάξαμε κυρίως, κυρίως ε, να δούμε πώς θα συνεργαστούν διάφορες κοινότητες. Συνήθως οι ερευνητές ε, λένε στους άλλους τι να κάνουν. Εμείς είπαμε ότι δεν πρέπει να γίνει έτσι. Πρέπει μεν να εμπνέουν τους δε. Έπειτα, οι χώρες έχουν η κάθε μία τη δική της δυνατότητα παρέμβασης, ε, το δικό της δυναμικό. Θα πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε όλα αυτά. Μετά από 3,5 χρόνια περίπου, μετά από αυτή τη διαδικασία, ε, φτιάξαμε ένα σχέδιο εφαρμογής που τρέχει ακόμα. Είπαμε λοιπόν, ας ε, ετοιμάσουμε δύο εργαστήρια συνδεδεμένα. Το πρώτο, φανταστείτε ότι έχετε ε, ένα πρόβλημα, ε, την προσωμίση του προβλήματος και αντιμετωπίστε το στο πρώτο εργαστήρι. Και στο δεύτερο, πώς μπορεί να συνεισφέρει η ερευνητική κοινότητα. Κάναμε λοιπόν στην, ε, ένα εργαστήρι στην Βαρσοβία και ένα εργαστήρι στη Ρώμη με διάφορους συμμετέχοντες, θέλω να πω σε λεπτομέρειες, συγγνώμη, στο Όσλο. Ε, στο Όσλο κάναμε ε, προσωμείωση του προβλήματος και είπαμε, ας πούμε, ότι δεν είναι, ε, ας πούμε, επίγον πρόβλημα. Αν θέλω ας πούμε, να περάσει ένα καλώδιο, αν, θέλει, ας πούμε, ε, αν θέλω να στήσω μία ανεμογεννήτρια, τι, γίνεται. Ε, σε αυτή την περίπτωση πρέπει να δούμε και το πρόβλημα των επενδύσεων. Ε, αν ε, θέλετε να παρακολουθήσετε μεγάλες εκτάσεις, είναι τόσο ακριβό αυτό το πράγμα. Ε, τιμάσαμε λοιπόν τέσσερις ομάδες, ε, την ομάδα διαχείρισης για το πώς ε, προσεγγίζει το πρόβλημα, το πώς ε, ανοιχνεύει και ταξινομεί τον κίνδυνο, τους, τους κινδύνους που μπορείς να προβλέψεις και την τεχνολογία που πρέπει να χρησιμοποιήσεις. Υπήρξαν πολλά επιστημονικά κενά. Τελικά φτάσαμε σε ένα κατάλογο, ε, καλέσαμε τους operators και καλέσαμε και τους επιστήμονες και φυσικά ποτέ δεν πάει το πράγμα όπως θα θέλαμε ιδανικά. Στο στη Ρώμη τι είπαμε. Ε, επειδή δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε όλα τα προβλήματα, ας εστιαστούμε στις προτεραιότητες και ας βάλουμε και νέες ιδέες. Δεν θέλουμε να προσεγγίσουμε απομονωμένα τα θέματα αυτά. Έχουμε την τεχνολογία, ε, τη διαχείριση ε, πρέπει να δούμε τα εργαλεία για τη λήψη των αποφάσεων. Γιατί πάντα πρέπει να βρούμε το συμβασμό ανάμεσα στο χρόνο και το χρήμα που χρειαζόμαστε. Είχαμε τέσσερις συνεδριάσεις. Ε, είδαμε τα εργαλεία για τις αποφάσεις, την χρήση της ε, τεχνητής νοημοσύνης, γιατί θέλαμε να μειώσουμε το κόστος παρέμβασης, οτιδήποτε σχετίζεται με τα χημικά και έπειτα ε, θέλαμε να βρούμε ευθυνούς τρόπους για να αντιμετωπίσουμε τις εκρήξεις. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες. Ε, όλα αυτά τα στοιχεία μπορείτε να τα πάρετε, να τα βρείτε, εν πάση σε κάθε μία από αυτέ τι συνεδριάσει ε, εντοπίστηκαν και ακούστηκαν πολλά πράγματα που μπορούν να, να γίνουν με διαφορετικές επενδύσεις. Ε, κάποια πράγματα ήταν πολύ εύκολα, ε, χρειάζονταν λίγα χρήματα κτλ. Κάποια περισσότερο. Το συμπέρασμα ποιο είναι. Ποια είναι η προσθέμενη αξία αυτή σε σχέση με το σημερινό σενάριο. Καταρχάς, έχουμε μια διαρθωμένη συνεργασία ανάμεσα στους επιστήμονες που μπορούν να προλάβουν και να ψάξουν να ερευνήσουν το πρόβλημα και τους operators. Έπειτα φτιάξαμε ένα ε, ήπιο πίνακο, όπως λέμε, soft table. Ε, οι επιστήμονες ε, είναι σε ένα απομονωμένο περιβάλλον και ασχολούνται με διαδικασίες μόνο. Τους δώσαμε λοιπόν αυτόν τον πίνακα για να ανταλλάσσουν πρακτικές ε, χωρίς να αγγίζουν τα κρίσιμα πράγματα και βάλαμε και το, την ιδέα του κόστους και του χρόνου και πώς θα εξοικονομήσουμε αυτούς τους δύο πόρους, κόστος και, χρόνος, και χρόνο. Λοιπόν, οι σκέψεις που προέγγιψαν. Συνήθως ε, το θεωρούμε αυτό ε, περιφερειακό πρόβλημα. Έχουμε στη Βαλτική, ας πούμε, ε, στην, ε, στο Βέλγιο, στη θάλασσα του Βελγίου, στην Ιταλία, ας πούμε, θεωρείται ότι είναι περιφερειακό το πρόβλημα. Έχουμε χώρους όπου πετάμε τέτοια ε, προϊόντα. Αλλά δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε απομονωμένα αυτό το πρόβλημα, ούτε γεωγραφικά, ούτε και κοινότητε. Δεν αφορά μόνο τι συγκεκριμένε κοινότητε. Και α υποθέσουμε ότι υπάρχει μία ε, κατεπίγουσα κατάσταση. Στην πραγματικότητα αντιμετωπίζουμε μόνο ε, βραχυπρόθεσμα αυτές τις κατεπίγουσες καταστάσεις. Και μετά το ξεχνάμε. Δεν θέλουμε να το αντιμετωπίζουμε όμω έτσι. Ε, θέλουμε να έχουμε μια προσέγγιση που θα συνδέεται και με το... θα έχει και χωρική διάσταση, αλλά ε, πιο συνολική ε, για το πώς θα αντιμετωπίσουμε ένα περίπλοκο πρόβλημα που συνδέεται με την, και με την νομοθεσία. Ξοδέψαμε δυόμιση χρόνια για να δούμε τι μορφή θα πάρει η συνεργασία για να καταλάβουν οι διάφορε κοινότητε η ε, μεν της δε και να εστιάσουν στις προτεραιότητες. Τους επόμενους τρεις τι ε, ετοιμάζουμε το συγκεκριμένο σχέδιο εφαρμογή, τα κράτη-μέλη και οι οργανώσει που χρηματοδοτούν την προσπάθεια βλέπουν τι προτεραιότητε έχουν και τι μπορούν να κάνουν. Θα ετοιμαστεί λοιπόν αυτό το σχέδιο εφαρμογής όταν τα κράτη-μέλη δουν τι δεσμεύσει ε, έχουν αναλάβει συνολικά και τι χρηματοδότηση διαθέτουν. μια και έχουμε λίγες ε, χρηματοδοτικές ευκαιρίες, δεν μπορούμε να τα καλύψουμε όλα. Ε, θέλουμε να δούμε την σκοπιμότητα, την ευρωπαϊκή προσθέμενη αξία και την ε, επίπτωση που έχει αυτή η προσπάθεια. Έχουμε πολλές ε, τεχνολογίες, μερικές είναι πολύ, πολύ ακριβές, μερικές δεν είναι πολύ γνωστές. Ε, εξετάσαμε όλες αυτές τις πτυχές. Αυτά. Ευχαριστώ. Thank Σας ευχαριστώ πολύ. Λέω να βάλω την αγγλική καμπίνα να δουλέψει λίγο και θα τα πω γερμανικά. Σας ευχαριστώ πολύ για τις παρουσιάσεις σας, αμφότερους. Όγγεν, έχεις κάποια ερώτηση? Δεν έχετε ακτή, έτσι, εδώ και παρκετό καιρό, εκεί κάτω. Ναι. Εγώ προέρχομαι από χώρα που δεν βρέχεται από θάλασσα, από την Αυστρία και με μεγάλο ενδιαφέρον άκουσα τα όσα είχατε να μας πείτε. Θα επανέλθω σε μία από τις πρώτες φράσεις που η κυρία Ράμος ανέφερε. Ότι δηλαδή 400.000 τόνοι χημικών όπλων βρίσκονται ποντισμένα στην Βαλτική θάλασσα. και ήλπιζα και ότι η επόμενη φράση θα ήταν από αυτούς τους τόνους έχουμε συλλέξει 450.000 τόνους. Αλλά δεν το άκουσα αυτό. 80 χρόνια μετά από τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο σχεδόν έχουν περάσει ε, και δεν έχει γίνει τίποτα. Δεν υπήρξε ευαισθητοποίηση, δεν υπήρχαν αρκετά κονδύλια. Τι έφτεξε. Επίσης, εκπλήσωμε και επομένως φτάνω στη δεύτερη ερώτησή μου. 21 χώρες έχουν εμπλακεί σε αυτήν την έρευνα. αλλά βλέποντας τα όσα συμβαίνουν και στη χώρα μου και σε άλλες χώρες, ε, διαπιστώνω ότι δεν συμμετέχουμε και αναρωτιέμαι το γεγονός ότι δεν έχουμε πρόσβαση στη θάλασσα σημαίνει ότι δεν ε, έχουμε καμία πραγματογνωμοσύνη για τα περί της ε, θαλάσσης. Ε, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν σπουδάσει και σχετικά θέματα και άλλωστε και στην Βιέννη υπάρχει και το Ινστιτούτο Θαλασσιών Μελετών. Αλλά ούτε και η Λετωνία δεν συμμετέχει. Αλλά βλέποντας το χάρτη Πραγματικά με εκπλήσει το γεγονός αυτό. Και το ερώτημα είναι ο αγωγός Nord Stream που είναι περίπου παράλληλος ε, με την ε, γραμμή καταβήθησης χημικών όπλων, έτσι όπως είδαμε σε μια διαφάνεια. Αυτό ε, ε, δημιουργεί κάποια προβλήματα σε σχέση με το North Stream. Σας είπε ποτέ κανείς ε, από τους υπευθύνου ότι α, βρήκαμε το τάδε ή το δίνα όπλο, βοηθήστε μας να το ανασύρουμε στην επιφάνεια. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Θα πω ότι πάνω σε αυτή την ερώτηση έχω να προσθέσω ότι υπάρχει μια δυσκολία στο να γνωρίζουμε ακριβώς πού ε, βρίσκεται τι. Και το σημαντικό είναι αυτοί οι χάρτες να είναι προσβάσιμοι σε όλους. έτσι ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα πληροφόρησης. Γι' αυτό λοιπόν ε, θα προσθέσω και εγώ στην ερώτηση του Όγγεν Φρόιντ και θα ρωτήσω το εξή, ότι ναι μεν έχουμε σχέδιο δράσης, όμως αυτό το σχέδιο δράσης δεν χρειάζεται συνεχόμενη δουλειά, επεξεργασία έτσι ώστε να επικαιροποιείται, να προστίθενται διάφορε δραστηριότητε, όπω για παράδειγμα η αγωγή που ανέφερε ο Γκεν Φρόιντ, έτσι ώστε να συμπληρώνεται το σχέδιο με τα αναγκαία στοιχεία. Ιδιαίτερα στην περίπτωση που υπάρχει βόμβα, πρέπει να αποσυναρμολογηθεί κομμάτι-κομμάτι και πρέπει ας πούμε να ε, απομακρυνθεί το νερό γύρω από τη βόμβα, πρέπει να προσέξουν πάρα πολύ οι πυροτεχνουργοί. Χρειάζεται να γίνουν πάρα πολλά και από πλευράς διοικητικής μέρημνας ε, και από πλευράς ασφάλειας, γιατί είναι επικίνδυνο. Γι' αυτό λοιπόν οι ειδικοί, η επιστήμη, η τεχνολογία, η πολιτική δεν θα έπρεπε να απαιτήσουν να προσθεθεί και ένα στοιχείο που να προβλέπει αυτόν ακριβώς τον καθαρισμό του βυθού. Εσείς τι έχετε να πείτε, ποια είναι η στάση της ε, αυτό και τι συμβαίνει με το διεθνές δίκαιο. Μπορούν όσοι το επιθυμούν να ξεκινήσουν δουλειά σε αυτό ή πρέπει να ακολουθήσουν διαφορετικές διαδικασίε, ε, να συμφωνήσουν με τους γείτονε α πούμε κτλ. Ε, να βρουν ποιοι έριξαν αυτά τα πολεμοφόδια και να αποδώσουν ευθύνε. Μπορούν ας πούμε ρώσικα πολεμοφόδια να απομακρυνθούν από άλλους. Πώς είναι τα πράγματα. Και Τι χρήματα υπάρχουν διαθέσιμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να γίνει κάτι τέτοιο. Υπάρχει κονδύλιο ή το μόνο που υπάρχει είναι τεχνική υποστήριξη και δεδομένα και τέτοια βοήθεια προς τα κράτη-μέλη. Διότι το οικονομικό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα. Γι' αυτό λοιπόν η Κομισιόν συνεισφέρει οικονομικά ή είναι μόνο συντονιστικός ο ρόλος της. Όγγεν, έχεις και άλλες ερωτήσεις ή όχι. Εσεί είστε από τη Λετωνία, άρα από τη μόνη χώρα που δεν συμμετέχει. Ξέρετε γιατί. Ε, thank you very much. Ε, Σας ευχαριστώ πολύ. Τις επιστημονικές λεπτομέρειες θα τις αφήσω στον συνάδελφο που ξέρει πολύ περισσότερα. Άρα Εξ όσων γνωρίζω και σε σχέση και με τη διαδικασία που προσπαθούμε να ολοκληρώσουμε τώρα, μπορώ να πω τα εξή. Ε, η στενή συνεργασία είναι κατά την άποψή μου το κλειδί, ε, κυρίως γιατί ε, αυξάνει την πίεση των ομοτήμων και δίνει κίνητρα στα κράτη-μέλη. για να κατανοήσουν ότι εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να ε, γίνει κάτι. Όσον αφορά την ε, ε, απόσυρση, την αφαίρεση, κοιτάξτε, πρόκειται για ένα πάρα πολύ λεπτό ζήτημα. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις υπάρχουν κύλινδροι των οποίων η αφαίρεση είναι πάρα πολύ δύσκολη ακόμα και αν τεχνικός ε, είναι εφικτή, ε, μπορεί να ε, μην γίνεται για άλλους λόγους. Ας πούμε, στην βελγική ακτογραμμή θα μπορούσε εύκολα να αφαιρεθεί ο κύλινδρος αλλά δεν είναι δυνατόν μετά να εξουδετερώσουμε τα αέρια τα οποία θα εκλειθούν. Προσπαθούμε να βλέπουμε κάθε φορά το θέμα από πολλές ε, σκοπιές και μέσα από περιφερειακά προγράμματα. Ας πούμε ε, υπάρχει η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Βαλτική, συγκεκριμένη δηλαδή στρατηγική για την ε, περιφέρεια αυτή, στρατηγική η οποία έχει προωθήσει αρκετά προγράμματα. Επίσης εμείς έχουμε δημοσιοποιήσει ε, μία, έναν διαγωνισμό υποβολής ε, προτάσεων όπου ζητούμε συγκεκριμένα projects που θα αντιμετωπίζουν αυτά τα συγκεκριμένα ε, προβλήματα. Γενικώ προσπαθούμε να ενθαρρύνουμε και τους εαυτούς μας και την βιομηχανία και τα κράτη-μέλη να επενδύσουν σε συστήματα τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση τέτοιων προκλήσεων. Ας πούμε, στο Horizon Europe αναφέρουμε ότι τέτοιου είδους προβλήματα πρέπει να απαντηθούν. Επίσης από πλευράς υποστήριξης και επενδύσεων και εκεί ζητούμε ε, κάποια υποστήριξη. Δυστυχώς πάντως πρόκειται για ένα πολύ λεπτό ζήτημα το οποίο χρειάζεται και τη βοήθεια της επιστημονικής κοινότητας φυσικά, αλλά και την βοήθεια από άποψη πολιτικού σχεδιασμού. Ε, υπάρχει και ειδική ομάδα στα πλαίσια της θαλάσσιας στρατηγικής ε, με, εντός του προγράμματος μέχρι το 2021 που ε, ασχολούνται και με το θέμα αυτό. Αυτό σημαίνει ότι βεβαίως θα εξαρτώμεθα και από την καλή θέληση των κρατών μελών, αν θέλουμε να έχουμε μια πραγματικά ε, συνολική προσέγγιση των θαλασσίων ε, σχεδιασμών. Όσον αφορά τώρα τις διασυνδέσεις και τους αγωγούς, είχαμε την περίπτωση του ε, Baltic Connector, που αναγκάστηκαν ε, να ε, κάνουν κάποια ιδιαίτερα χρονοβόρα αλλά ε, και ακριβή μετακίνηση της σχεδιασμένης γραμμής ακριβώς γιατί βρήκαν πυρομαχικά. Οπωσδήποτε ο θαλάσσιος χώρος ε, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με ιδιαίτερο ε, τρόπο έτσι ώστε να μην προκύψει κίνδυνος ούτε για τους πληθυσμούς ούτε για το περιβάλλον. Ευχαριστώ. Υπάρχουν δύο σχόλια τα οποία απολύτως ευθυγραμμίζονται με τις ερωτήσεις που συνήθως ε, δεχόμαστε. Να ξεκαθαρίσουμε λοιπόν πρώτα απ' όλα δύο πεδία γιατί δεν έχουν απομακρυνθεί και δεύτερο γιατί δεν ε, συμμετέχουν κάποιες χώρες όπως ε, η Αυστρία. Γιατί λοιπόν ε, δεν προχωρούμε σε απομάκρυνση. λόγω χρημάτων και λόγω προτεραιοτήτων αν θέλω να είμαι πολύ απλός. Και μετά τεχνικές ε, ε, ικανότητες ε, επίλυσης των προβλημάτων αυτών. Τα προβλήματα αυτά μέχρι τώρα έχουν αντιμετωπιστεί, έχουν θεωρηθεί ως, ως προβλήματα που αφορούν τις χώρες και τα εδάφη τους. Οι υπηρεσίες οι οποίες είναι υπεύθυνε ε, για να αντιμετωπίσουν έκτακτες καταστάσεις ξέρουν πάρα πολύ καλά πώς να τις αντιμετωπίσουν. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ε, ε, ε, το να πέσει κανείς ε, πάνω σε μια βόμβα ας πούμε και να πρέπει να την απομακρύνει, να την εξουδετερώσει και μια, και μια μεγάλη παρουσία τέτοιων αντικειμένων σε ευρεία θαλάσσια περιοχή. Αυτό είναι τελείως διαφορετικό πρόβλημα και εδώ αυτό είναι το, η μεγάλη πρόκληση. Το ζήτημα είναι πώς να εκτιμήσει και να αξιολογήσει καλές, ε, κανείς διαφορετικές ε, ε, επιλογές ή εναλλακτικές. Ανάλογα με την παρέμβαση που πρέπει να κάνεις, πρέπει να κάνεις και τη σωστή επιλογή. Η δικιά μας υπηρεσία αυτό που κάνει είναι να, κάνει, να προσεγγίζει το θέμα μέσα από πολλαπλές μελέτες επιπτώσεων οικολογικών, περιβαλλοντικών, οικονομικών κλπ. Και βεβαίω το, το ζητούμενο είναι να βρει κανεί ε, τις εναλλακτικέ που έχει. Και υπάρχουν και εναλλακτικέ οι οποίες είναι πολύ δύσκολο να τις διαχειριστεί κανείς. Στην ε, JPC Oceans ε, συμμετέχουν και χώρες που έχουν πρόβλημα και άλλες που δεν έχουν άμεση, άμεσο πρόβλημα. Πάντως η συμβολή της επιστημονικής κοινότητας που μπορεί να είναι ε, ε, μια συμβολή μεμονωμένου ε, ερευνητή ή κάτι πολύ πιο ευρύ μας οδηγούν στο να θέσουμε και προτεραιότητες. Αλλά στο τέλος της ημέρας το ζήτημα είναι να δούμε ποιο είναι το αποτέλεσμα και το αποτέλεσμα θα πρέπει να είναι διαθέσιμο σε όλους. Τέλος, είπατε τι γίνεται με ανταλλαγή καλών πρακτικών. Σε επιστημονικό επίπεδο αυτό γίνεται ούτως ή άλλως μεταξύ επιστημόνων. Ε, μερικές φορές ε, μπορεί να ε, υπάρχουν κάποιοι δισταγμοί, αλλά σε γενικές γραμμές ε, είναι Ε, ε, είναι κοινή πρακτική. Απ' την άλλη πλευρά ε, υπάρχουν ας πούμε πεδία γνωστικά τα οποία εξ αρχής δεν θεωρούσαν ότι μπορούν να συμβάλλουν. Ας πούμε κοινωνικοί επιστήμονες τους οποίους εμείς βάλαμε στο παιχνίδι τώρα μέχρι κάποια στιγμή θεωρούσαν ότι δεν μπορούν να συμβάλλουν στην λύση τέτοιου, τέτοιων προβλημάτων. Δεύτερον, η πρόσβαση ε, των δεδομένων, όχι σε επίπεδο επιστημονικής κοινότητας. Δηλαδή, στοιχεία τα οποία πρέπει να, στα οποία πρέπει να έχουν πρόσβαση οι αρμόδιες αρχές. Μπορεί να βρεθούν στο διαδίκτυο. Είναι πάντως ένα μείγμα ανάμεσα σε δημόσια πρόσβαση ή ε, πρόσβαση κατά το μάλλον ή τον ελεύθερη. Ε, το ζήτημα είναι λοιπόν ποιος έχει την ιδιοκτησία των δεδομένων στα οποία πρέπει να υπάρχει πρόσβαση. Ξέρετε, το θέμα αυτών των πυρομαχικών δεν διαφέρει και πολύ από άλλα προβλήματα, είτε διατροφικά είτε άλλα. Uh, Θα ήθελα λοιπόν να κάνω μια συγκεκριμένη ερώτηση για το North Stream. Γιατί είναι πάρα πολύ κοντά στο κέντρο του προβλήματος. Έχουν γίνει κάποιες κινήσεις για να βοηθήσουν τους ε, κατοίκους εκεί με το πρόβλημα, για το πρόβλημα αυτό. Στην περίπτωση μας, δεν μπαίνουμε σε λεπτομέρειες ε, όταν γίνεται ένα συγκεκριμένο αίτημα, διότι υπάρχουν αρμόδιες αρχές. Αυτό που κάνουμε είναι να εξετάζουμε το πώς η επιστήμη και η τεχνολογία μπορούν να συνεισφέρουν και πώς να μειωθεί το κόστος της παρέμβασης. Εάν λοιπόν η αρχή που είναι αρμόδια είναι μια τοπική, μια παγκόσμια αρχή, είναι κάποια βιομηχανία όμως, γιατί μπορεί πολλές φορές ε, μια βιομηχανία να αναλαμβάνει την απομάκρυνση πολεμοφοδίων για να προστατέψει ένα καλώδιο που έχει περάσει, για παράδειγμα. Εξαρτάται από την κάθε περίπτωση. Ε, δεν ξέρω να σας πω αυτή τη στιγμή. Μπορούμε όμως να ρωτήσουμε, να μάθουμε. Ναι, αλλά μπορεί όμως να έχουν και οι ίδιοι εθνικοί ασποφορείς ή οποιοδήποτε άλλοι εμπειρογνώμονες που είναι κάνει να ε, χειριστούν αυτά τα πολυμοφόδια. Ναι, να σας απαντήσω. Υπάρχουν ενδελεχείς μελέτες που έχουν γίνει και που γίνονται προτού ξεκινήσει μια τέτοια διαδικασία Γι' αυτό και είναι τόσο σημαντική η χαρτογράφηση. Και πιστεύω ότι τόσο ε, στον Αρκτικό ωκεανό τόσο και στην ε, Βαλτική είναι πάρα πολύ σημαντική η χαρτογράφηση. Νομίζω πως ε, η κατάσταση στη Μεσόγειο είναι καλύτερη, βέβαια δεν είναι ιδανική. Γι' αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντική η χαρτογράφηση. Όταν έχεις τις λεπτομέρειες και γνωρίζεις πού βρίσκονται αυτά τα πολεμοφόδια, είναι πολύ πιο εύκολο να τα απομακρύνεις. Αλλά υπάρχει μια περίπτωση πριν από ένα μήνα, α πούμε, που στη Βόρεια Θάλασσα ένα πλοίο χρειάστηκε να αλλάξει πορεία γιατί ε, υπήρχαν τέτοια καταβυθισμένα πολεμοφόδια στη ρότα του. Δεν έχουμε λάβει έτοιμα από το North Stream για ε, να παρέχουμε βοήθεια, ακριβώς επειδή έχουν τους δικούς τους ε, εμπειρογνώμονες και ειδικού. Ναι, αλλά οι χάρτες όμως είναι διαθέσιμοι σε όλους. Δεν είναι στρατιωτικό απόρριτο ή μυστικό, α πούμε. Αν κάποιο βρει ένα χάρτη δεν τον κρατήσει για τον εαυτό του. Υπάρχει μια γενικότερη συμφωνία για να είναι προσβάσιμοι σε όλους οι χάρτες αυτοί. Ναι, για έργα όπω αυτό, οι κυβερνήσει των κρατών μελών δίνουν πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα όταν εγκρίνουν ένα τέτοιο πρόγραμμα απομάκρυνση. Όμως σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν υπάρχει ακόμα κάποιο εργαλείο που να συνδυάζει όλες αυτές τις πληροφορίες και να τι παρουσιάζει μαζί. Γι' αυτό χρειάζεται να δοθεί πολιτική προσοχή ακριβώ επειδή ναι μεν η επιστήμη είναι ε, εκεί παρούσα αλλά χρειάζεται και πολιτική βούληση και γι' αυτό εμείς έχουμε το σχέδιο δράσης ε, για την θάλασσα στο οποίο αναφέρεται η ανάγκη συντονισμένης προσέγγισης έτσι ώστε να έχουμε μια ιδέα του τι έχουμε και τι δεν έχουμε, τι, τι μπορούμε να κάνουμε, πού βρίσκεται το καθετή. Σας ευχαριστώ. Νομίζω πως αυτή ήταν μια ικανοποιητική απάντηση. Να προσθέσετε κάτι. Να σας πω ότι οι χάρτες είναι πάρα πολύ σημαντικοί. Γιατί, Γιατί δεν είναι στατικά, στατικά αυτά τα ε, πολεμοφόδια. Μετακινούνται, ξέρετε, με τα ρεύματα. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να επικαιροποιούνται Επίση, η Βαλτική δεν είναι το ίδιο με τη Μεσόγειο, υπάρχει άλλο βάθος, οπότε και άλλες δραστηριότητες χρειάζονται για να απομακρυνθούν. Χρειάζεται λοιπόν να εντοπίσουμε τις προκλήσεις και να τις αντιμετωπίσουμε, διότι όταν έχεις ένα αντικείμενο που το ψάχνει μηχάνημα, ε, έχεις να κάνεις με, την, με προβλήματα εντοπισμού. Είτε αυτό είναι αρχαιολογικό έβριμα, είτε αυτό είναι πολεμοφόδιο. Χρειάζεται λοιπόν και τεχνολογική γνώση και από την άλλη είναι και θέμα ε, φυσικής κιόλα, το πώς κυκλοφορούν τα ρεύματα, πώς αλλάζει ο βυθός της θάλασσας. Ο χάρτης λοιπόν ε, που δείχνει την τοποθεσία δεν σου δείχνει και απαραίτητα το που βρίσκεται ο κίνδυνος. Ωραία, ευχαριστώ μπορώ να τολμήσω ένα πολιτικό συμπέρασμα και να πω ότι φυσικά όταν υπάρχει διαθέσιμη πληροφορία πρέπει αυτή να είναι προσβάσιμη και όταν αλλάζει κάτι, δηλαδή όταν εξουδετερώνεται ένα τέτοιο, ένας τέτοιος κίνδυνος, χρειάζεται να επικαιροποιούνται και οι χάρτες. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται ένας μηχανισμός που να προβλέπει αυτές τις ε, διαδικασίες και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να δημιουργήσει ένα πρόγραμμα που να συλλέγει όλες αυτές τις πληροφορίες και να τις συνδυάζει. Ίσως ε, να μην είναι απαραίτητα συντονιστικό πρόγραμμα τα κράτη-μέλη, αλλά ενημερωτικό. Έτσι ώστε όλοι οι φορείς που θέλουν να αναλάβουν τέτοιες δραστηριότητες μάκρυνες πολεμοφοδίων να γνωρίζουν με τι έχουν να κάνουν και πώς έχει κατάσταση. Εφόσον λοιπόν δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις ή σχόλια από τους συναδέλφους, θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήρθατε σήμερα. Να σας ευχηθώ καλή συνέχεια και ελπίζω να καταφέρετε τους στόχους σας. Με τη βοήθειά μας ίσως. Uh, Συνάδελφοι, το επόμενο θέμα έχει προγραμματιστεί για τις 10.30, οπότε να σας ενημερώσω πώς θα κάνουμε ένα διάλειμμα 35 λεπτών, έτσι ώστε να κάνετε και εσείς διάφορες δουλειές. Επιστρέψτε όμως 10.30. Okay, dear colleague. <laughs> Αγαπητοί συνάδελφοι, resume our meeting and uh, we, we Ξαναρχίζουμε λοιπόν τη συνεδρίασή μα, σημείο 13 τη ημερησίας διατάξεως, προοπτικέ τυποποίηση των εξοπλισμών σε Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ. Θα ανταλλάξουμε απόψεις λοιπόν με τον κύριο Εβάρντας, Μαζέικης ε, εδώ το έγραψε λάθος αλλά εγώ επειδή έχω feeling ε, με την λιθουανική γλώσσα και τα ξέρω αυτά είπα θα έχουμε μετά τον κύριο Χαράλαμπο Γιανακόπουλο από τη Γενική Διεύθυνση Grow Και θα έχουμε και τον Τζον Γιάνσεν, πρόεδρο της Συμβουλευτικής Ομάδας Επιτεχνικών Θεμάτων του ΝΑΤΟ και ανώτερο σύμβουλο για θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ίδρυμα Βιομηχανικών Άμυνας και Ασφάλειας των Κάτω Χωρών. Η συζήτησή μας νομίζω ότι είναι πάρα πολύ, ότι έρχεται την κατάλληλη στιγμή γιατί και η ΕΝΤΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση ασχολούνται πολύ με τα θέματα αυτά. Ελπίζουμε ότι και με το σχετικό ταμείο θα έχουμε το, ε, τα κονδύλια τα οποία θα μας επιτρέψουν την αναμενόμενη τυποποίηση με ε, προθεσμία λίγο μακρινή όσον αφορά το MFF ε, θα δούμε ε, και είναι η κατάλληλη ώρα να δούμε ποιες είναι οι ικανότητες που έχουν η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Άμυνας και τι μπορούμε να κάνουμε έτσι ώστε να βοηθήσουμε την τυποποίηση. Είχαμε ήδη μία πρώτη ανταλλαγή απόψεων ε, κατά την ε, παρουσίαση της την, την παρουσίαση της μελέτης θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Μαζέικης πρώτα. Ευχαριστώ πολύ. Έχω 10 λεπτά, έτσι δεν είναι. Ναι, βέβαια, έχετε 10 λεπτά. Πρώτα απ' όλα, ε, χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ, παρότι η αίθουσα δεν είναι γεμάτη. Ε, ε χαίρομαι Είμαι αναπληρωτή ε, διευθυντή Διεύθυνση Βιομηχανία Συνεργειών και Καταρρυτικών Παραγόντων ε, στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνα. Η τυποποίηση ε, είναι πραγματικά σημαντική σε τον τομέα. Πριν φτάσω στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνα, ήμουν στην υπηρεσία τυποποίησης του ΝΑΤΟ για πολλά χρόνια και ίσως να είμαι αυτός που μπορεί να συνδυάσει με πολύ καλό τρόπο ε, τους δύο αυτούς κόσμους ας πούμε. Ε, γνωρίζω πάρα πολύ καλά πώς λειτουργούν τα, τα πρότυπα και ε, ξέρω και τι γίνεται πλέον και με τα πρότυπα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς αντιμετωπίζουμε τα πρότυπα. Από εκεί να ξεκινήσουμε η δική μας προσέγγιση όσο γίνεται λιγότερο μη στρατιωτική και μόνο τα χρειάζεται στρατιωτική. Ε, θέλουμε ε, μη στρατιωτικά πρότυπα ε, σε πολλούς ε, χώρους και σε πολλά πεδία. Ο τρόπος λειτουργίας ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, διαφέρει βέβαια από τον τρόπο λειτουργίας του ΝΑΤΟ. Προσπαθούμε να συμμετάσχουμε ε, στους οργανισμούς ανάπτυξης τυποποίησης που μπορούν να επηρεάσουν την δημιουργία των πρωτοτύπων από την πρώτη στιγμή και με τρόπο ώστε να γίνουν πλέον καταλληλότερα για την δική μας αμυντική βιομηχανία. Υπάρχει Eurocire που αφορά τα πρότυπα ε, της ε, αεροπλοείας ε, και συμμετέχουμε λοιπόν και σε αυτή τη διαδικασία και συμμετέχουμε επίσης και με το δικό μας input έτσι ώστε τα πρότυπα να λειτουργήσουν σωστά και προς όφελός μας. Αυτό είναι ένα γενικό πλαίσιο για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τα πρότυπα. Δεν δημιουργούμε όμως πρότυπα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς διευκολύνουμε και προσπαθούμε να βοηθήσουμε τις αμυντικές κοινότητες, κοινότητες να επιτύχουν τα πρότυπα. Αλλά ε, αν θέλουμε τα ε, πρότυπα θα πρέπει να σταθούμε προς τη Sense Electing έτσι κλπ. Ε, μπορούμε να στραφούμε επίσης και στο ΝΑΤΟ και να δούμε ε, ε, αυτά τα πρότυπα τα οποία εκεί έχουν ήδη δημιουργηθεί. Οι κύριες δραστηριότητες τις οποίες έχουμε πλέον στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνα. Να σας πω ότι πέρσι εγκρίναμε τη στρατηγική ευρωπαϊκής τυποποίησης για την άμυνα. Είναι η πρώτη φορά που έχουμε ένα τέτοιο έγγραφο το οποίο προσπαθεί ε, να διευθετήσει όλες τις διαδικασίες οι οποίες ε, αποσκοπούν εις την τυποποίηση των εξοπλισμών ε, και έχει επιφέρει και πολλές βελτιώσεις στην διαδικασία διαχείρισης προτύπων και τυποποίησης. Μια δεύτερη φάση είναι η PFMP Πρόκειται για το Project Standardization ε, Plan. Θέλουμε να αντιμετωπίσουμε τα θέματα της τυποποίησης ήδη από την δημιουργία του project. Ε, ξεκινώντας ένα project πρέπει να ελέγξουμε ε, αν υπάρχουν ήδη πρότυπα διαθέσιμα, ή αν υπάρχουν κενά, ποιος θα πληρώσει τα ελλειπή πρότυπα κτλ είναι μια διαβίου κατά κάποιο τρόπο διαδικασία η οποία ακολουθεί το project σε όλη τη διάρκεια ζωής του. Υπάρχει και η ENEU, το PSNP, εργαλείο το οποίο εγκρίναμε πρόσφατα, πέρσι συγκεκριμένα, και τώρα έχουμε κάποια πιλωτικά δοκιμαστικά προγράμματα όπου προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό το εργαλείο το οποίο θα το βελτιώνουμε σιγά σιγά. Αυτά τα δύο πιλωτικά ε, είναι η ERPAS και Single Open Sky. Πρόκειται για δύο ε, σημαντικά ε, προγράμματα για, τον, για την EDA. Ναι, ναι, και αυτά ε, συμμετέχουν ε, στα drones. Έχουμε και την ε, Ιάζα όμως η οποία ασχολείται περισσότερο με αυτά. βέβαια να σας πω ότι ένα drone μου κάνανε και μένα δώρο, το βρήκα κάτω από το χριστουγεννιάτικο δέντρο, αλλά εδώ μιλάμε για άλλου είδους ε, drones. Μιλάμε για άνοιγμα φτερών 20 μέτρων. Ε, αυτά για το Airpass, αλλά τώρα να γυρίσω στην τυποποίηση. Θα πρέπει να δούμε και ποια είναι τα σημεία στα οποία μπορούμε να βελτιώσουμε ε, την διαδικασία. Ξέρετε ότι έχουμε αυτή τη δεύτερη γενιά προγραμμάτων 35 προγράμματα συγκεκριμένα και πρέπει να τα ελέγξουμε και από τη σκοπιά της τυποποίησης. Αν θέλουμε τα προγράμματα να είναι επιτυχή, θα πρέπει να δούμε από την αρχή την διαλειτουργικότητα. Ε, μια ικανότητα η οποία δεν έχει τη δυνατότητα ε, ε διαλειτουργικότητας ε, δεν θα προχωρήσει καλά. Εμείς ε, αλλάξαμε λίγο τα ονόματα της Γενικής Διευθύνσης, της Διευθύνσης στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άνμινας. Ε, να σας πω ότι πριν, όταν έπρεπε να πω ποιος είμαι, ε, έπρεπε να δώσω ένα πάρα πολύ μακρύ τίτλο ενώ τώρα μπορώ να πω ότι είμαι στη διεύθυνση συνεργειών και καταλυτικών παραγόντων critical enablers. Είναι πιο εύκολο και για μένα. Αυτό ε, προέρχεται από την ευρωπαϊκή στρατηγική, αλλά να σας πω ότι οι καταλητικοί παράγοντες ε, αφορούν ε, και τον εξοπλισμό και τα πρότυπα και είναι ένα από τα κεντρικά στοιχεία εάν θέλουμε να επιτύχουμε συνολική αυτονομία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και βεβαίως ε, είναι γεγονός ότι δεν μπορούμε να ελέγξουμε όλους τους εξοπλισμούς ε, ταυτόχρονα. Ε, γι' αυτό είναι καλό πράγμα η τυποποίηση. Βλέπω ότι έχει περάσει, έχουν σχεδόν περάσει τα 10 μου λεπτά και πρέπει να εξάγω κάποια συμπεράσματα. Κατά την άποψή μου ως εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας, είναι σημαντικό να πούμε μερικά πράγματα. Είναι σημαντικό να χρησιμοποιήσουμε τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας σαν σημείο εισόδου για τις διαδικασίες τυποποίησης. Όντως, ε, εάν δείτε ε, όλα τα υφιστάμενα ε, θεσμικά όργανα κτλ. Ε, θα δείτε ότι στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας έχουμε διεύθυνση που ασχολείται με την τυποποίηση, έχουμε ε, διεύθυνση η οποία ασχολείται με τα European Standard Reference. Επίσης εκεί ε, περιλαμβάνεται και κατάλογος με τις βέλτιστες πρακτικές όσον αφορά την τυποποίηση και γενικώ πιστεύω ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας είναι το καλύτερο φόρουμ για την ε, διαχείριση των προτύπων των εξοπλισμών. Ε, στο ε, έγγραφο το οποίο ανέφερα προηγουμένω, είναι πολύ βασική σημασία όσον αφορά την τυποποίηση σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση και χαίρομαι που ο Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας αναφέρει το εξής. Ε, η Κομισιόν πρότεινε στην ε, ε, ΕΟΑ να ξεκινήσει ένα σχέδιο δράσης για την τυποποίηση σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Τυποποίησης και πιστεύω ότι όταν θα έχουμε υλοποιήσει την ευρωπαϊκή πολιτική τυποποίηση της άμυνας θα έχουμε ανταποκριθεί σε, αυτό το, σε αυτή τη δουλειά και σε αυτό το καθήκον. Αυτά και αν θέλετε είμαι στη διάθεσή σας και αν μου το επιτρέψει ο Πρόεδρος να απαντήσω και στις ερωτήσεις σας. Επόμενος είναι ο κύριος Γιανακόπουλος. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ που με καλέσατε να μιλήσω για αυτό το σημαντικό θέμα. Όπως είπε και ο προηγούμενος ομιλητής, Δουλεύω στη Γενική Διεθνήση Grow ε, στο δεύτερο τμήμα που ασχολείται με την άμυνα και θυμάμαι γιατί είμαι αρκετό χρόνο εκεί, ε, πώς ξεκίνησε και πώς εξελίχθηκε η αμυντική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2013 μέχρι σήμερα. Το 2013 η τυποποίηση ήταν ένα από τα βασικά σημεία της ανακοίνωσης του 2013 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ήταν η πρώτη σημαντική ανακοίνωση για την άμυνα και το 2014 επίσης το θέμα της τυποποίησης υπήρχε και ήδη από το 2013 είπαμε πως τι δράσεις θα πρέπει να προωθήσουμε για να βελτιώσουμε τις πολιτικές το τομέα της τυποποίησης των αμυντικών συστημάτων. Δύο ήταν οι βασικοί λόγοι. Ο πρώτος είναι προφανής. Αυτές οι βελτιώσεις, την τυποποίηση θα μπορούσαν και θα έπρεπε να οδηγήσουν στην καλύτερη διαλειτουργικότητα των αμυντικών συστημάτων για τις ευρωπαϊκές Αναπλές δυνάμεις. Αυτός ήταν ο απότατος σκοπός. Να μπορούμε δηλαδή να πηγαίνουμε σε επιχειρήσεις και να επιχειρούμε μαζί με άλλες νατοικές δυνάμεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, χωρίς προβλήματα, απρόσκοπτα, σε όλες τις δυνατότητες από το επιμελητιακό μέχρι τις πραγματικές επιχειρήσεις. Αυτό είναι το ζητούμενο. Ο άλλος στόχος είναι να μειώσουμε το κόστος. Φυσικά είναι πολύ σημαντικό αυτό, να μειώσουμε το κόστος σε όλες τις δραστηριότητες των ενόπλων δυνάμεων. Από την κατάρτιση, απόκτηση εξοπλισμού, συντήρηση του εξοπλισμού, ε, και για να ανοίξουν και οι αμυντικές αγορές, οι αγορές αμυντικών εξοπλισμών. Με τη χρήση όλο και περισσότερο κοινών προτύπων στα συστήματα που χρησιμοποιούμε και που αγοράζουν οι ένοπλες δυνάμεις. Αυτό θα, οδηγούσε σε μια, θα οδηγήσει σε μια λιγότερο κατακαιρματισμένη αγορά. Και αυτό έχει πολλά πλέον εκτήματα. Δηλαδή, αν έχεις ε, κοινές, κοινά πρότυπα, κοινά, κοινές στρατηγικές ε, στα συστήματα, έχεις την, ίδια, την ίδια αρχιτεκτονική, μπορείς να ανοίξεις τις ε, αγορές, σε πολλές εταιρείε, μπορείς να αυξήσεις τις πιθανότητες να βρεις ε, ε, ανταλλακτικά εξαρτήματα λοιπά από παντού σε όλο τον κύκλο ζωής των ε, εξοπλισμών σου. Αυξάνεις τον ανταγωνισμό, αυξάνεις την αγορά σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν και θα έχουν πρόσβαση σε υποσυστήματα ή εξαρτήματα των εξοπλισμών σου. Θα, θα πέσει το κόστος φυσικά γιατί ο ανταγωνισμός θα μειώσει το κόστος και θα έχουμε λιγότερες επικαλύψεις βεβαίως. Μια ανοιχτή αγορά δίνει ευκαιρίες και μπορείς να έχεις πολλές εναλλακτικέ λύσεις στη διάθεσή σου. Επομένως, ε, μπορεί να, οδηγήσει, μπορεί να οδηγήσει σε πιο ενιαία αγορά, λιγότερο κατακαιρματισμένη, με περισσότερες ευκαιρίες για όλους σε όλη την Ευρώπη. Το πρόβλημα είναι πώς θα το πετύχεις αυτό. Και ποιες είναι οι βασικές τάσεις που υπάρχουν στον χώρο. Υπάρχουν πολλές δραστηριότητες για να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, να αυξήσουμε, να προωθήσουμε τη χρήση των κοινών προτύπων και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας μπορεί να παίξει κάποιο ρόλο εδώ, ε, μπορεί να βοηθήσει την απλούστευση των διαδικασιών και βεβαίως και το ΝΑΤΟ να παίξει το ρόλο του. Υπάρχουν βεβαίως διάφορες παράμετροι που επηρεάζουν ε, τα δεδομένα ε, και δεν έχουν να κάνουν το αμυντικό, με την αμυντική βιομηχανία. Έχει να κάνει με το μη στρατιωτικό επίπεδο. Υπάρχει όλο και μεγαλύτερη χρήση ε, μη στρατιωτικής ε, τεχνολογίας στον αμυντικό τομέα. Και αυτό ε, σημαίνει ότι και τα πρότυπα που χρησιμοποιούνται στο μη στρατιωτικό τομέα ε, τα χρησιμοποιεί και θα πρέπει να μπορεί να τα χρησιμοποιεί και ο αμυντικός κλάδος η μη στρατιωτική τεχνολογία ε, και οι εξελίξεις ε, αφορούν όλο και περισσότερο το στρατιωτικό επίπεδο. Και η ανάπτυξη προτύπων σε αυτούς τους ε, τομείς θα επηρεάσουν και τον τομέα της άμυνας και θα δημιουργήσουν μία πιο ενιαία τελικά χρήση των προτύπων και στον τομέα της άμυνας. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα μη στρατιωτικά πρότυπα αρκούν για τον αμυντικό κλάδο. Υπάρχουν προσαρμογές, πρέπει να γίνουν σε ορισμένε φάσεις ε, προσαρμογές και επίσης θα πρέπει να δούμε σε ποια φάση της δημιουργίας των ε, προτύπων ε, για, την μη για το μη στρατιωτικό κλάδο θα πρέπει να εμπλακεί ο στρατιωτικός, το επίπεδο, το αμυντικό επίπεδο για να ληφθούν υπόψη οι δικές του ανάγκες. Μια άλλη τάση που υπάρχει και θα δούμε πώς θα επηρεάσει τη χρήση κοινών προτύπων είναι μια τάση που υπάρχει όλο και μεγαλύτερη και που προσπαθούμε να την προωθήσουμε με τις δράσεις μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Κομισιόν είναι να φτιάχνουμε και να σχεδιάζουμε ε, από κοινού διάφορα αμυντικά συστήματα με τη συμμετοχή διαφορών χωρών. Αν έχουμε κοινά project για τις τοπικές δυνατότητες μας, είναι υποχρεωτικό να χρησιμοποιούμε τα ίδια πρότυπα για τα ίδια συστήματα. Τμήμα, από, τμήμα των, του κατακαιρματισμού που βλέπουμε στα πρότυπα οφείλεται στο γεγονός ότι έχουμε πολλαπλά προγράμματα και συστήματα στην Ευρώπη. Όσο προωθούνται τα προγράμματα συνεργασίας, θα δούμε ότι μειώνεται η ανάπτυξη διαφορετικών συστημάτων στην Ευρώπη και επομένως ε, μειώνεται και η χρήση διαφορετικών προτύπων και τα, τα πρότυπα θα γίνονται όλο και πιο κοινά. Θα προωθούνται τα κοινά πρότυπα στην Ευρώπη όλο και περισσότερο. Κάτι άλλο τώρα. Θα ήθελα να σκεφτούμε, να δούμε πότε... Πρέπει να δούμε πότε σκεφτόμαστε τη δημιουργία προτύπων ε, για την ανάπτυξη συστημάτων. Κάποια στιγμή στο ερευνητικό επίπεδο, όταν φτάσουμε όταν, ε, στη φάση της έρευνας, το σκεφτόμαστε. Δεν θα πρέπει να το κάνουμε πολύ νωρί, γιατί η έρευνα δεν αφορά την τυποποίηση της τεχνολογίας, είναι να βρει νέα πράγματα, να πειραματιστεί με νέα πράγματα, να σκεφτεί εφάνταστα και όχι να επαναλαμβάνει τα ίδια μοντέλα και σχήματα. Κάποια στιγμή όμως οι τεχνολογίες οριμάζουν και τα συστήματα πηγαίνουν προς, την, προς τον τελικό σχεδιασμό και τότε θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τα πρότυπα. Αυτό το κάνουμε ήδη. Και το τμήμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ασχολείται με την έρευνα, με τις προπαρασκευαστικές του δράσεις για τον αμυντικό τομέα, αλλά ακόμα και πιο πριν στα πιλωτικά προγράμματα Από τη στιγμή που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είπε ότι πρέπει να υπάρχουν πιλωτικά προγράμματα, υπάρχουν project τα οποία αφορούν ε, τα, την διαλειτουργικότητα των συστημάτων και είχαμε ένα πιλωτικό πρόγραμμα, ε, το Strava, για τις διαδικασίες στην παρασκευαστική δράση το 2017 αφορούσε μια αρχιτεκτονική ε, με ανοιχτά πρότυπα για, τους... για συστήματα που τα χρησιμοποιούν οι στρατιώτες. Το 2019 έχουμε ένα άλλο πρόγραμμα που δεν έχει δημοσιευτεί. Θα υπάρξει ένα project, ένα ειδικό project για την τυποποίηση και τη λειτουργικότητα. Επιπλέον, πέρα από αυτά τα project, στο διαγωνισμό του 2018 είχαμε φτάσει αρκετά υψηλό επίπεδο ρημότητας. Προσπαθήσαμε να δούμε τις προϋποθέσεις για τα πρότυπα. Και οι προϋποθέσεις είναι να χρησιμοποιούμε όσο δυνατόν περισσότερο τα ισχύοντα πρότυπα και να ε, σεβόμαστε και τα πρότυπα του ΝΑΤΟ όσο μπορούμε περισσότερο μερικές φορές να κάνουμε συγκεκριμένη αφορά ε, σε συγκεκριμένα, συγκεκριμένους αριθμούς προτύπων, το τάδε πρότυπο δηλαδή, ε, με αυτόν τον τρόπο η αγορά θα είναι λιγότερο κατακαιρματισμένη, θα πλουστευτεί και η προσπάθεια της, της έρευνας των ερευνητών για να φτάσουμε σε κάτι το οποίο να είναι χρήσιμο και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί κιόλα από πολύ περισσότερους χρήστες. Με αυτό το πιο συγκεκριμένο τρόπο μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα με ρεαλιστικό τρόπο. Τώρα, δεν ξέρω τι εξέλιξη θα υπάρξει. Όπως σας είπα, η δημιουργία και η υιοθέτηση προτύπων είναι εθελοντική. Δεν ε, την επιβάλλουμε σε κανέναν και δεν θα έπρεπε να επιβάλλεται σε κανέναν. Ακολουθεί τη λογική της αγοράς. το γιατί έχουμε κατακαιρματισμένες αγορές, υπάρχουν λόγοι και πάντα είναι οι ίδιοι λόγοι. Όσο θα χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο μη στρατιωτική τεχνολογία και όσο θα έχουμε περισσότερα συνεργατικά προγράμματα στην Ένωση, βαθμία, θα βλέπουμε μια πιο ενιαία προσέγγιση απέναντι στα πρότυπα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. And next is... Ευχαριστούμε. Επόμενος ομιλητής ο κύριος Γιάνντσεν. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Αγαπητά μέλη της Επιτροπής, σήμερα στην παρουσίασή μου θα ασχοληθώ με δύο στοιχεία. Πρώτα θα σας εξηγήσω τη θέση και το ρόλο της ε, Συμβουλευτικής Ομάδας Τεχνικών Θεμάτων του ΝΑΤΟ και έπειτα θα σας ε, πω δύο λόγια για την τυποποίηση γενικότερα ε, με τον κύριο Τζοβάνι Ρωμάνη συνεργαστήκαμε για αυτήν την παρουσίαση. Ο κύριος Τζοβάνι είναι υπεύθυνο για θέματα τυποποίηση στο ΝΑΤΟ. Όπως γνωρίζετε, 22 μέλη του ΝΑΤΟ είναι και μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τον λόγο αυτό, οι σχέσεις ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πάρα πολύ σημαντικές. Αν υπολογίσουμε και τους εταίρους διαλειτουργικότητας όπως ονομάζονται, ο αριθμός ε, των ε, συνεργατών λοιπόν αυξάνεται και ε, ενέρχεται σε 25 από συνολικά 28 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε κοινέ αξίες. Και θα έλεγα ότι έχουμε και μια κοινή βάση φορολογούμενων πολιτών και αυτό είναι εξίσου σημαντικό διότι σημαίνει ότι τα χρήματα των φορολογούμενων θα πρέπει να δαπανώνται με τρόπο όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερο. Η Συμβουλευτική Ομάδα Επιτεχνικών Θεμάτων του ΝΑΤΟ συμμετέχει στην ε, ΣΥΝΕΤ, την ε, Ομάδα Διευθυντών για Θέματα Άμυνας από τις ε, δηλώσεις του ΝΑΤΟ βλέπουμε ότι είναι πολύ σημαντική η πρόθεση της συνεργασίας. Και να σας ε, παρουσιάσω τον τρόπο λειτουργίας του ΝΑΙΑΓ, της Συμβουλευτικής Ομάδας ε, του ΝΑΤΟ. Πρώτον, είναι, ένας, είναι μια ομάδα που υπάγεται στο ΝΑΤΟ. και δεν είναι εξωτερική συμβουλευτική ομάδα ούτε λόμπι. Και παρά το γεγονός ότι υπόκειται στο CNET, είμαστε στη θέση να βοηθήσουμε οποιαδήποτε άλλη υποομάδα ή οργανισμό που υπάγεται στο ΝΑΤΟ. Βρισκόμαστε σε συνεγή ανταλλαγή πληροφοριών με την Ευρωπαϊκή Ένωση και οι συμβουλές που παρέχουμε είναι στο πλαίσιο των ε, μη ανταγωνιστικών δραστηριοτήτων του ΝΑΤΟ. Εμείς ε, δεν ε, θέλουμε να εισέλθουμε σε κάποια σύγκρουση συμφερόντων. Δεν μας ενδιαφέρει κάτι τέτοιο. Μας ενδιαφέρουν θέματα διαλειτουργικότητας, στις στην οποία διαλειτουργικό, η διαλειτουργικότητα μάλλον είναι κάτι στο οποίο μπορούν να συμμετέχουν ε, όσοι το επιθυμούν. Σε γενικές γραμμές ε, περνάνε τρία χρόνια από μια αρχική έκθεση μέχρι το αποτέλεσμα. Έχουμε λοιπόν μια αρκετά εκτεταμένη εργαλειοθήκη που παρέχει συμβουλές ε, στους ενδιαφερόμενους. Τώρα, η διάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν υπάρχει τόσο καλή οργάνωση όσο στο ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση, η e UMS και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουν αυξήσει τις προσπάθειες για βελτίωση της, συνεργασίας, της αμυντικής συνεργασίας. Οι δομές λοιπόν εξελίσσονται και αυτές με ε, δυναμικό τρόπο. Και νομίζω πως θα συμφωνήσετε όλοι ότι ο στόχος για τον εξοπλισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι οι ε, δαπάνες με πιο συνετό τρόπο. Θα πρέπει να υιοθετηθεί μια ολιστική προσέγγιση. Και αυτό που λείπει αυτή τη στιγμή από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η βιομηχανική διάσταση από όλες τις δραστηριότητες που έχουν σχέση με ε, οπλισμό. Χρειάζεται λοιπόν να καλυφθούν αυτές οι ελλείψεις διότι πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε σε θέση να παρέχουμε συμβουλές και βοήθεια σε όσους το ζητούν. Οι αμυντικές ικανότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να είναι συμβατές με την ε, διαλειτουργικότητα και να ακολουθούν τις τεχνολογικές εξελίξεις. Το Ινστιτούτο Στρατηγικών Σπουδών ε, με επικεφαλή τον κύριο Ντανιέλ Φιότ έχει εκδώσει μία μελέτη σχετικά η οποία είναι εξαιρετική και στην έκθεση αυτή αναφέρεται σε ό,τι φορά την ΝΑΙΑΚ ότι η οδηγία για τον οπλισμό δεν προβλέπει άμεση υποβολή εκθέσεων αλλά πρώτερη διαβούλευση. Τα κράτη λοιπόν είναι εκείνα που αποφασίζουν και όχι η βιομηχανία. Μετά, τα πρότυπα αναπτύσσονται για διαφορετικούς λόγους στην κάθε περίπτωση. Στην ε, μη στρατιωτική αγορά χρησιμοποιούνται εξαιτίας ε, της ε, ζήτησης της ίδιας της αγοράς. Για παράδειγμα το USB το ξέρετε όλοι, το χρησιμοποιείτε όλοι. Ο κυριότερο στόχο λοιπόν είναι η διαλειτουργικότητα. Επίτευξη διαλειτουργικότητα μαζί με. Ε, σε όλα τα κράτη. Για παράδειγμα, βελληνικές. Ο συνάδελφός μου από την Εθνική Υπηρεσία Άμυνας σίγουρα μπορεί να σας πει και περισσότερες ε, λεπτομέρειες για αυτό και για το πόσο σημαντικό είναι. Τώρα, ε, ήταν το Στάνεκ επιτυχημένο εγχείρημα. Θα μπορούσε, εάν τα κρατημέλη όχι μόνο είχαν κυρώσει την ε, συμφωνία, αλλά και την είχαν εφαρμόσει. Η εφαρμογή του Στάνεκ σε ένα συγκεκριμένο project πρέπει να συνδυαστεί και με ρεαλιστικούς στόχους και με τις ε, πραγματικές ε, δυνατότητες ε, της κάθε χώρας. Σε περίπτωση που αυξάνεται το κόστος υπερβολικά, τότε τα κράτη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μια πιο οικονομική επιλογή. Το 2019 το πρόγραμμα που έχει σχεδιαστεί απαιτεί διαλειτουργικότητα σε ό,τι αφορά τον οπλισμό και η βιομηχανία οφείλει να τηρήσει αυτήν την ε, προϋπόθεση. Η οικονομία επίσης καθορίζει τα πρότυπα. Η βιομηχανία παράγει πρότυπα τα οποία δεν εξυπηρετούν όλους τους σκοπούς της ε, διαλειτουργικής άμυνας κατά ανάγκη. Ακόμα και αν δημιουργούνται πρότυπα εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν είναι υποχρεωτικό να είναι συμβατά με τις απαιτήσεις που έχει το ΝΑΤΟ. Και δημιουργείται έτσι ε, κίνδυνος να μην εφαρμόζονται αυτά τα πρότυπα. Ε, ωστόσο, αν ξεκινήσει η διαδικασία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχει κίνδυνος να μην είναι συμβατή σε περιβάλλον ΝΑΤΟ. Η ιδανικότερη λοιπόν λύση θα ήταν μια προσέγγιση κατά περίπτωση. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ και θα παρακολουθήσω τη συζήτηση με μεγάλο ενδιαφέρον. Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω τώρα το λόγο στους συναδέλφους. Ποιος έχει ερώτηση, κύριε Στρογεύσκη. Θα μιλήσω πολωνικά. Βάλτε τα ακουστικά σας λοιπόν. Θα ήθελα ευθύς εξ αρχής να πω το εξής. Και μην το πάρετε προσωπικά. Ε, δεν αισθάνομαι ικανοποιημένο και λίγο απογοητευμένο. Γιατί από την αρχή της κοινοβουλευτικής θητείας Ακούγαμε τις εξής πληροφορίες, ότι η τυποποίηση και κάποιοι, κάποια πρότυπα σε ό,τι αφορά την ασφάλεια ε, συνεπιφέρουν κάποιες, έχουν κάποια αξία. Όταν έχεις πρότυπα, αυτό είναι σημαντικό. Αλλά όμως είναι εθελοντικά και πρέπει πάρα πολλά να γίνουν ακόμα αυτά τα έχουμε ξανακούσει, μας τα έχουν ξαναπεί, τα ξέρουμε. Αλλά το πιο σημαντικό είναι το εξής. Θα ήθελα να μου πείτε αυτή η διαδικασία τι μορφή παίρνει ε, και πώς εξελίσσεται για τις διάφορες ομάδες συμφερόντων. Δεν έχουμε όλες τις πληροφορίες. Φερρυπίν για, για την άμυνα. Ας πάρουμε τις μεταφορές, την κινητικότητα, την επιμελητία. Σε αυτούς τους τομείς Όλοι λένε ότι το να βάλουμε πρότυπα σημαίνει ότι είμαστε πιο αποτελεσματικοί και μειώνεται το κόστος ε, για τις μεταφορές. Μιλάω για τις στρατιωτικές μεταφορές και τις μεταφορές που συνδέονται με, το με τον τομέα της, βιομηχα... της άμυνας. Το θέμα είναι τι πρόοδος έχει συμβεί σε αυτόν τον τομέα. Έπειτα, ε, ανεπάνδρωτες λύσεις, όπως τα drones, ανεπάνδρωτα οχήματα, αεροπλάνα και ελικόπτερα. Υπάρχουν κάποιες, κάποιοι κανονισμοί σχετικά που όμως δεν έχουν προχωρήσει πολύ. Κάποια κράτη-μέλη θέλουν κανονισμούς για την ασφάλεια των drones, ειδικά όταν χρησιμοποιούνται από ιδιώτες για ιδιωτικούς, ιδιωτικούς σκοπούς. Μιλάμε για τη χρήση τους από ανθρώπους που δεν έχουν καμία σχέση με το αμυντικό κλάδο. Αλλά παρόλα αυτά μπορεί η επιρροή τους να είναι πολύ σημαντική. Ε, το Ηνωμένο Βασίλειο έκαναν κάτι σχετικό, η Γαλλία και η Γερμανία για την ασφάλεια των drones. Έχουμε δηλαδή δέσμες ε, κανόνων και κανονισμών που δεν είναι όμως ε, συνεπεί και δεν κινούνται όλοι προ την ίδια κατεύθυνση. Από τη μία μιλάμε τόσο πολύ για την τυποποίηση, αλλά όμω αυτό το συγκεκριμένο τομέα αυτό που συμβαίνει είναι αποσπασματικές λύσει και, λύσεις και σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει μια, ένας μονόδρομος. Πολλές, πολλές χώρες μιλάνε ε, για το θέμα και τον τομέα της πολιτικής αεροπορίας. Δεν θέλουν να μείνουν παθητικές σε, αυτές τις, σε αυτόν τον τομέα. Θα πρέπει ίσως να παρέπετε περισσότερο εσείς, ούτω ώστε να εξασφαλιστεί αυτή η συνέπεια που θέλουμε ε, όλοι μας Φαρμακοβιομηχανία επίσης. Η φαρμακοβιομηχανία ε, έχει διάφορα εμπορικά project και, και αυτά έχουν πολλά προβλήματα γιατί ο καθένας κάνει τα δικά του. Δεν υπάρχει κανένα ενιαίο πρότυπο. Ίσως λοιπόν θα πρέπει να κάνουμε πολύ περισσότερα και σε αυτό το επίπεδο. Ακόμα και για εκπαιδευτικούς σκοπούς, για το καλό της κοινωνίας μας, για να αποφύγουμε πιθανούς κινδύνους και απειλές. Χρειαζόμαστε επίσης τυποποίηση στη, στα κανάλια επικοινωνίας. Εγώ έχω ακούσει πολλούς ομιλητές να έρχονται εδώ και να λένε ότι κάποια κανάλια επικοινωνίας αλληλοεπικαλύπτονται, ότι δεν υπάρχουν πρότυπα για τον τρόπο επικοινωνίας μας γενικώ, ότι υπάρχουν πάρα πολλές απειλές που δεν αναλύονται επαρκώς, γιατί δεν υπάρχει ένα κεντρικό σημείο, ένα κομβικό σημείο που να συγκεντρώνει τις πληροφορίες, να συγκεντρώνει την πραγματογνωμοσύνη και να μας επιτρέπει να αντιδράσουμε αποτελεσματικά. Λόγω του γεγονότος ότι δεν έχουμε τυποποιημένα κανάλια επικοινωνίας, ότι δεν έχουμε έναν μονοσήμαντο ορισμό για τα επίπεδα απειλής. Μπορούμε να έχουμε πληροφορίες που από κάποιους μπορούν να θεωρούνται ασήμαντες, να αγνοούνται και ως αποτέλεσμα να είμαστε πιο αδύναμοι αντί για πιο δυνατοί. Επίσης, ποια είναι η πρόοδος που έχει σημειωθεί σε ό,τι αφορά την τυποποίηση στους τομείς που σας ανέφερα. Καλό θα ήταν να μας δώσετε συγκεκριμένα παραδείγματα για να μας πείτε πού πάνε καλά τα πράγματα της τυποποίησης, σε ποιο κλάδο, πού υπάρχουν ε, αντιδράσεις, πού δεν προχωράει το πράγμα. Είμαι πεπισμένος ότι σε πολλούς τομείς ε, η τυποποίηση που έχει προσθέμενη αξία θα πρέπει να είναι ο στόχος μας για να είμαστε πιο αποτελεσματικοί, να βελτιώσουμε το επιμελητιακό επίπεδο και να μειώσουμε το κόστος. Σημαντικό. Ευχαριστώ. Άλλες ερωτήσεις από τους άλλους συναδέλφους. Όχι. Στον κύριο Γιάντσεν, μια και μας συστήσατε ότι το ισοδύναμο του ΝΑΙΑΚ θα πρέπει να υπάρχει και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ΝΑΙΑΚ αποτελείται από βιομηχάνους από τις χώρες του ΝΑΤΟ. Οι περισσότερες χώρες όμως είναι και μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα έχει νόημα λοιπόν να ανοίξετε τον ΆΙΑΚ. Δηλαδή να έχουμε ε, αυτούς ε, τους ανθρώπους, αυτούς τους βιομήχανους είναι από τη Σουηδία, ε, Φιλανδία, Ιρλανδία και Αυστρία. Για να έχουμε τα ίδια πρότυπα σε Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ. Γιατί καλό θα ήταν να έχουμε τα ίδια όπλα, ας πούμε, όλοι. Δεν θα έχει νόημα λοιπόν ε, οι ίδιοι πάνω κάτω άνθρωποι να έχουν τις ίδιες πληροφορίες και στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποιος θέλει να απαντήσει τις ε, παρατηρήσεις του Ευρωβουλευτή μας από την Πολωνία με την ίδια σειρά. Μπορείτε να ξεκινήσετε λοιπόν να απαντάτε με την ίδια σειρά. Σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Δεν ήταν ερώτηση, είχε και σχόλιο μέσα κύριε Ζρογεύσκη αλλά νομίζω πως ε, τονίσατε τη, τους σημαντικούς τομείς της τυποποίησης. Ίσως δεν θα μπορέσω να καλύψω όλα τα κομμάτια της ερώτησής σας, αλλά μας ρωτήσατε για την πρόοδο που έχει σημειωθεί σε κάποιους τομείς όπως ε, στα μη επανδρομένα οχήματα, όπως για παράδειγμα τα drones. Υπάρχουν διάφοροι κανονισμοί, υπάρχουν διάφοροι φορείς που ε, εμπλέκονται, η Άσα καταρχάς ε, που προσπαθεί να αναρμονίσει ε, την νομοθεσία με τα drones. Τα drones αυτή τη στιγμή είναι περίπου, είναι στις εκατοντάδες χιλιάδες, αλλά μέχρι του χρόνου θα έχουν φτάσει στα εκατομμύρια. Η, η Άσα λοιπόν είναι ένας φορέας, μετά η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Άμυνας, η προσπαθούμε να εκπροσωπούνται όλοι οι φορείς άμυνας. Επίσης, Eurokai, που ασχολείται με πρότυπα στην αεροπορία και με μεγαλύτερα μη επανδρομένα οχήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για στρατιωτικούς σκοπούς. Μετά υπάρχει η ομάδα συντονισμού και τυποποίησης UAS ε, για μη επανδρομένων ε, οχημάτων δηλαδή. Η ομάδα αυτή προσπαθεί να ασκήσει επιρροή στη διαδικασία τυποποίησης έτσι ώστε να οδηγηθούμε σε παγκόσμια πρότυπα. και υβριδικά πρότυπα. Μετά, πάμε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και εδώ θα δούμε ότι στο ΝΑΤΟ οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός εταίρος με εξαιρετικά αναπτυγμένο σύστημα drones. Εκεί υπάρχει το Τζάρος, είναι ένα διεθνές φόρουμ τυποποίησης το οποίο ασχολείται ιδιαίτερα με τα συστήματα και το λογισμικό αυτών των μη επανδρομένων οχημάτων. Σε αυτό το επίπεδο λοιπόν προσπαθούμε να φέρουμε σε επαφή και τις δύο πλευρές, ε, Ευρώπη και Αμερική. Όμως χρειάζεται να παρακολουθούμε τις εξελίξεις, γιατί είναι πολύ σημαντικό για μας να υπάρχουν πρότυπα τόσο για τα drones όσο και γενικότερα για τα μη επανδρομένα οχήματα. Επίσης, ε, υπάρχει μια νέα μορφή σκάφου στο λεγόμενο mail, μέσω ύψος μακράς ε, διάρκειας, το οποίο χρειάζεται επίσης τυποποίηση γιατί είναι κάτι καινούργιο. Το ΝΑΤΟ επίσης χρησιμοποιεί το σύστημα AGS. Και οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ έχουν ήδη επενδύσει πολλά σε αυτό το σύστημα, όμως ε, ακόμα υπάρχουν ελλείψεις σε ό,τι αφορά την τυποποίηση. Τώρα, υπάρχουν διάφορες διακλαδώσεις μεταξύ αυτών. Το Τζάρος είναι αμερικανικό, το ΙΑΣΑ ασχολείται και με μη στρατιωτικά θέματα. Υπάρχει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Άμυνας. Προσπαθούμε λοιπόν να φέρουμε όλους αυτούς τους οργανισμούς στο τραπέζι και να συνεργαστούμε. Τώρα, αναφερθήκατε και στην στρατιωτική κινητικότητα. Αυτό είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα για να δούμε πώς μπορούμε να συνεργαστούμε με το ΝΑΤΟ και να βελτιωθούν τα πρότυπα ως αποτέλεσμα. Μπορούμε να εξετάσουμε, για παράδειγμα, αν όλα τα πρότυπα ε, είναι συμβατά με τη στρατιωτική κινητικότητα. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Άμυνας ασχολείται με αυτό το θέμα. Επίσης υπάρχει και το πρόγραμμα ΠΕΣΚΟ από... με την ε, συμμετοχή πολλών χωρών και έδρα της κατοχώρες. Τώρα, θα δώσω το λόγο στους συναδέλφους για να συνεχίσουν. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Γιανακόπουλε, θέλει να πείτε κάτι. Uh, I mean, we're not here for but I can... Δεν έχω απαντήσεις ίσως, αλλά μπορώ να σας δώσω ένα παράδειγμα. Συζητούσα πριν από καμιά δυο μέρες με εκείνους που ασχολούνται με το πρόγραμμα επίδειξης Οκεανός ε, 2020 ε, που εντάσσεται στις παρασκευαστικές δράσεις ε, πρέπει να γίνει μία επίδειξη στη Μεσόγειο και μία στη Βαλτική και στην επιδείξεις αυτές υπάρχουν επιχειρήσεις πολλών των συστημάτων που δραστηριοποιούνται στον ίδιο χώρο, στον ε, τάμενων εναέριων συστημάτων δηλαδή, και με ε, σταθερά πτερήγια και με περιφερ... Ε, ε που περιστρέφονται, περιστρεφόμενα. Δεν θα σας το περιγράψω περί, περίπου. Τα αριθμιστικά ε, οι ρυθμιστικέ πτυχέ που πρέπει να ληφθούν υπόψη, τόσο ότι αυτά τα πράγματα να μπορέσουν να συνεπάρξουν στον ίδιο χώρο. Είναι τόσο περίπλοκο αυτό. Μην φανταστείτε ότι είναι μόνο τα εναέρια που είναι περίπλοκα. Ε, μπορούμε να έχουμε και υποβρύχια ας πούμε, συστήματα στο λιμάνι. Πώ μπαίνουν στο λιμάνι, πώ βγαίνουν από το λιμάνι. Όλα αυτά είναι καινούρια και τα πλαίσια που έχουμε στην διάθεσή μας αυτή τη στιγμή δεν είναι επαρκή για αυτά τα νέα συστήματα. Πρέπει να βελτιώσουμε το ρυθμιστικό επίπεδο και να τυποποιήσουμε τα ρυθμιστικά συστήματα σε κάθε χώρα και για ένα, συστήματα τα οποία υπάρχουν ήδη, όπως ας πούμε τα ενάρια συστήματα, αλλά και τα ανεπάνδρωτα υποβρύχια ε, συστήματα ή συστήματα επιφανείας. Υπάρχουν οργανώσεις οι οποίες ε, κάνουν δουλειά, πρέπει να λυθούν υπόψη τα όσα έχουν κάνει. Δεν είναι απλό. Ε... Κατά τη διάρκεια αυτών των ασκήσεων, τουλάχιστον θέλουμε να δούμε ποια είναι τα προβλήματα. Ε, στο συγκεκριμένο project, αυτό που ρωτήσαμε και δεν προβλεπόταν στην αρχή ήταν να μας πούν οι ειδικοί λεπτομερώς ποια είναι τα αριθμιστικά και διοικητικά προβλήματα, ούτως ώστε αυτά τα συστήματα να μπορούν να συνεπάρχουν. Αν, γιατί αν για ένα γυμνάσιο, για μια επίδειξη, για ασκήσεις έχουμε προβλήματα, φανταστείτε τι γίνεται σε επιχειρήσει. Τα έχουμε πολύ περισσότερα. Δεν γίνεται. Φυσικά υπάρχουν λύσει ad hoc, υπάρχουν παρεκκλήσει, αλλά δεν μπορούμε να τα αφήσουμε με τι παρεκκλήσει όλα αυτά τα πράγματα να λειτουργούν στο μέλλον. όλες αυτές οι, ε, σε όλες αυτά τα επίπεδα συμμετέχουν πολλοί, πολλοί φορείς. Θυμάμαι το 2013 ε, θέλαμε να ετοιμάσουμε ένα πλαίσιο για τα εναέρια συστήματα, τόσο ώστε να ε, ενσωματωθούν ε, στο εναέριο χώρο μέχρι το 15-16 αυτά τα εναέρια συστήματα και έχουμε φτάσει στο 19 και ούτε κατά διάνοια δεν το έχουμε πετύχει. Επομένως είναι ένα νέο καθήκον. Ε, ψάχνουμε να βρούμε όλοι μας. Είναι πιο περίπλοκο από ό,τι είχαμε φανταστεί. Και είναι περίπλοκο γιατί είναι καινούριο. Γιος Γιάνσεν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν έχω συγκεκριμένη απάντηση όσον αφορά τα πρότυπα, αλλά όσον αφορά το σημείο το οποίο θίξατε, για ε, μέλη της ΕΝΑΙΑ που έρχονται από, την, ε, τα Ηνωμένα Έθνη και εξηγούν τι συμβαίνει και λαμβάνουν υπόψη το περιβάλλον του ΝΑΤΟ. Αυτό είναι κάτι το οποίο κατάλαβα στην αρχή της ε, θητείας μου. Γι' αυτό ορίσαμε στην ομάδα τον λεγόμενο EU Rapporteur έτσι ώστε να δίνει την άποψη του περιβάλλοντος άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εισηγητής της Ευρωπαϊκής Ένωσης δηλαδή. Για λόγους πληροφοριακούς ε, καταρχήν, για να δούμε λοιπόν με ποιο τρόπο μπορούμε να εξελίξουμε την βιομηχανική αμυντική συνεργασία. Ναι, είναι και αυτό ένα άλλο στοιχείο. Από την άλλη πλευρά, η ΝΑΙΑΚ ως σώμα του ΝΑΤΟ ε, λειτουργεί σύμφωνα με τις αρχές και 25 αποστολές ε, στο ΝΑΤΟ είναι μέλη και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μερικές φορές ε, μπορεί να εκφράσουν διαφορετική άποψη σε διάφορα φόρα. Και επομένως εμείς ως σώμα του ΝΑΤΟ θα πρέπει να, να βλέπουμε πάντα οτιδήποτε μας ε, ε, ζητάτε υπό τη σκοπιά του ΝΑΤΟ. Να σας πω επίσης ε, ότι δεν θα είμαστε και σε θέση να δώσουμε συγκεκριμένη παροχή συμβουλών για τα προγράμματα τα οποία προκύπτουν ίσως από την ΕΣΚΟ, ίσως από την EDA. Σας ευχαριστώ πολύ. Η ιδέα μου από τεχνικής απόψεως ήταν ε, να πάρουμε τους βιομηχάνους από, από αυτές τις χώρες ε, μέλη ε, για να συζητήσουν και με ανθρώπους που δεν είναι, με χώρες που δεν είναι στο ΝΑΤΟ. Αυτό που σκεφτόμουν να είναι το εξής, οι βιομηχανοί δεν μιλάνε με την ίδια γλώσσα και από τις δύο πλευρές ή ε, ενδεχομένως ε, οι δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι του ΝΑΤΟ μπορεί να πούνε κάτι άλλο από την ε, από ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι στην ίδια κυβέρνηση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά οι βιομηχανοί δεν έχουν τέτοιες εμπλοκές. Ξέρουν ποιο είναι το συμφέρον τους και ενδιαφέρονται γι' αυτό ανεξαρτήτως πλαισίου. Γι' αυτό έλεγα να υπάρχει κάποια εναρμόνιση των μέσων. Ωραία. Ολοκληρώσαμε λοιπόν αυτό το σημείο της ημερησίας διατάξεως. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους και βεβαίω όταν ξεκινήσει η νέα θητεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είμαι σίγουρο ότι ε, θα σα ξαναδεί αυτή η επιτροπή μια άλλη, με, με μια άλλη ευκαιρία. Ωραία. Το επόμενο σημείο τώρα τη ημερησία διατάξεω που είναι και το τελευταίο. Έπρεπε να ξεκινήσει στις 11.30 και 30 ε, και αφορά ενημέρωση σχετικά με την άσκηση Trident Juncture 18 και θα έχουμε μαζί μας τον ε, Αντινάμεχο και την Όλσεν στρατιωτικό εκπρόσωπο της Νορβηγίας στο ΝΑΤΟ και την Αλεσάνδρα Προκόπιο που είναι στο Διεθνές Προσωπικό Τμήμα Επιχειρήσεων του ΝΑΤΟ. Παρακαλώ πολύ ε, όλους όσοι δεν έχουν δικαίωμα να παραμείνουν στη συνεδρία και κλεισμένων των ε, θυρών ε, να εγκαταλείψουν την αίθουσα. Θα ξεκινήσουμε στις 11.30 ακριβώς.